περιμένουμε λοιπόν θετικέ εξελίξεις μετά από δύο άσχημα χρόνια. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Επίτροπε. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για τη Μαδαγασκάρη. Η ψηφοφορία θα γίνει περίπου σε μισή ώρα. Δεύτερο σημείο. Agenda is Guantanamo. Το επόμενο σημείο λοιπόν στην ημερήσια διάταξη είναι η επικείμενη απαγγελία θανατικής ποινής στο Γουαντάναμο. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τάνο, όπω και προηγουμένω. Κύριε Πρόεδρε, οι μεταρρυθμιστέ και οι συντηρητικοί θεωρούν ότι η θανατική ποινή είναι θέμα ε, συνείδησης για το αν θα είναι κανείς υπέρ αλλά δεν θα πρέπει να επιβάλλονται τέτοιες ποινές σε κάθε περίπτωση. Ε, παρόλο που έχουμε εκατομμύρια συμπολιτών μας που είναι υπέρ της θανατικής ποινής, εδώ μιλούμε για την πιθανότητα απαγγελίας θανατικής ποινής ε, εις βάρος πολύ επικίνδυνου τρομοκράτη που συνομωτούσε για την ε, δολοφονία χιλιάδων αθώων. Και μάλιστα ε, πριν από έξι χρόνια ζήσαμε και το τρομοκρατική επιθέση στο Λονδίνο, στην εκλογική μου περιφέρεια. Μερικές φορές ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας έχει ανα, απρόβλεπτα αποτελέσματα και η, ο χώρος κράτησης στο, στον κόλπο του Γαντάναμου αντικατοπτρίζει αυτή την τραγική κατάσταση και κυρίως ε, το δυσβάσταχτο βάρος και το ασύμετρο σχέση με τους υπόλοιπους που φέρουν οι Αμερικανοί στον αντιτρομοκρατικό αγώνα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια δημοκρατική χώρα, συμμεριζόμαστε τις ε, ίδιες αρχές. Βέβαια, οι τέτοιου είδου δίκες θα πρέπει να γίνονται με τις προδιαγραφές ε, του διεθνούς δικαίου και κατά προτίμηση από πολιτικά και όχι στρατιωτικά δικαστήρια. Κυρία Αναγκόμες η Ευρώπη ορθώνει το ανάστημά της κατά της ε, θανατικής ε, πηγής, ε, ποινής και θα πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί. Και η Λέδη και η επερχόμενη Πολωνική Προεδρία θα πρέπει να το επαναλάβουν. Η περίπτωση του Αλ Ραχίμ Αλ Νασίρη δεν είναι η μοναδική. Όμως, εάν του απαγγελθεί η θανατική ποινή, όχι μονάχα θα είναι κακό για τις ίδιες τις Πολιτείες, αλλά θα είναι και πολύ αρνητικό στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Ο πρόεδρος Ομπάμα δεν θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το κληροδότημα του πρόεδρου Μπούς όσον αφορά την καταπάτηση δικαιωμάτων ε, ε, στο όνομα της καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας. Τα οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει ε, και οφείλουν να κάνουν περισσότερα και εμείς ε, θα πρέπει ε, να τους πιέσουμε έτσι ώστε να αλλάξει η απόφαση αυτή. Επίσης να σταματήσουν τα στρατιωτικά δικαστήρια διότι δεν έχουν τις προδιαγραφές για δίκαιη δίκη και επίσης ε, να μην έχουν πλέον το δικαίωμα να κρατούν ε, φυλακισμένους ανθρώπους τους οποίους δεν έχουν απαγγελθεί ε, καταγγελίε. Ο Αλ Νασίρη εδώ και εννέα χρόνια είναι φυλακισμένος και ξέρουμε ότι έχει περάσει από μυστικό ανακριτικό κέντρο της CIA στην Πολωνία. Θα πρέπει να, δει, να δοθεί η δυνατότητα να βρει το δίκιο του όποιος έχει υποστηρίξει υποστεί βασανιστήρια και όποιος δεν έχει ε, δεχτεί μια δίκαιη δίκη ε, ενώπιον ε, στρατιωτικού δικαστηρίου. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως ισχύει και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κατσμάρεκ σήκωσε μπλε κάρτα. Τη δέχεστε κυρία Γκόμες. Κύριε Πρόεδρε, έχω μία ερώτηση προς την κυρία Γκόμες. Από πού έχετε την πληροφορία για μυστικές φυλακές της CIA στην Πολωνία. Δεν έχετε απόδειξη για τέτοιου ισχυρισμού. Μπορεί να έχετε εσεί τέτοιε αποδείξει, πληροφορίε από έγκυρε πηγέ, αλλά εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Εσεί από πού το ξέρετε, κυρία Γκόμε. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξήγαγε μια ε, έρευνα για το σύστημα παράνομων μεταγωγών και πήγαμε στην Πολωνία και σε δύο άλλες χώρες ε, για τις οποίες υπήρχαν ισχυρισμοί μυστικών φυλακών. Στην Πολωνία και την ε, Ρουμανία υπήρχαν υπόνοιες για μυστικές φυλακές και από ό,τι ξέρουμε κάτι συνέβη, κάτι βρέθηκε και στην Λιθουανία και μάλιστα ξεκίνησε κοινοβουλευτική έρευνα για το θέμα αυτό. Από την επερχόμενη Πολωνική Προεδρία το μόνο που περιμένουμε είναι να διεξαγάγει κανονική έρευνα προκειμένου να διαλευκανθεί το ζήτημα και να αποκατασταθεί η αλήθεια για αυτούς τους πολύ σοβαρούς ισχυρισμούς της βάρος της Πολωνίας. Βλέπω δύο ακόμη μπλε Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μπλε κάρτε σε απάντηση που ακούγεται σε προηγούμενη μπλε κάρτα, γιατί ήταν συνέχεια της προηγούμενη μπλε Κυρία Βερζιά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Γκουέ αποφάσισε να μην προσυπογράψει αυτό το ψήφισμα για το Γουαντάναμο. Δεν είμαστε κατά του ψηφίσματος, αλλά θεωρούμε ότι παρά είναι μετριοπαθές. Λυπούμε για τον τρόπο με τον οποίο εκπονήσαμε το ψήφισμα αυτό. Πολλές επιφυλάξεις, πολύ επιφυλακτικός τόνος για να καταδικάσουμε την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μια χώρα που υποτίθεται είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, που παρόλα αυτά εφαρμόζεται θανατική ποινή και μάλιστα το Γουαντάναμο δείχνει πώς η χώρα αυτή παραβιάζει ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα στο όνομα του αντιτρομοκρατικού αγώνα. Έχουμε έναν άνθρωπο που πάνω από 10 χρόνια βρίσκεται στο κουβανέζικο έδαφος σε αμερικανική βάση και μάλιστα θα καταδικαστεί ε, χωρίς, χωρίς καμία απόδειξη για πολλούς από αυτούς που κρατούνται στο Γουαντάναμο αυθαίρετα και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους κρατούμενους υπέστησαν βασανιστήρια ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος, στη Ρουμανία, τη Λετωνία, την Πολωνία, αλλά αυτά δεν πρέπει να τα λέμε γιατί πώ να δίνουμε μαθήματα και να κάνουμε κηρύγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα αν εμεί οι ίδιοι είμαστε ανίκανοι να τα σεβαστούμε στην επικράτειά μα. Και φυσικά δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο στο σημερινό ψήφισμα. Λυπούμε ειλικρινά, αλλά δεν πιστεύω ότι έτσι θα, θα προωθήσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόμμα. Φυσικά θα πρέπει να εμποδίσουμε τη θανατική καταδίκη του κυρίου Αμπτελ Ραχίμ Αλνασίρη και πολλών άλλων. Αλλά δεν μπορούμε να ε, απλώς να λυπούμαστε για την υπαναχώρηση του Προέδρου Ομπάμα σε ό,τι αφορά την ε, σύσταση στρατιωτικών δικαστηρίων. Μπλε κάρτα του κύριου Πρέντα. Do you accept the blue card? Mr. Preda, go ahead. Δέχεστε κύριε Βεζιάτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση προς την κυρία Βεργιά και λυπάμαι που δεν πρόλαβα να θέσω την ίδια ερώτηση πριν στην κυρία Γκόμες. Κυρία Βερζιά, πιστεύετε ότι ε, εξακοντίζοντα τέτοιε κατηγορίε κατά τη Ρουμανία αντίστοιχε με αυτέ τη κυρία Γκόμες κατά τη Πολωνία, πιστεύετε ότι έτσι θα βοηθήσετε την υπόθεση του κυρίου Αλνασίρη. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι οι κατηγορίες σας αυτές θα μας βοηθήσουν να βρούμε τρόπο για να αναχαιτήσουμε την απαγγελία θανατικής ποινή. Νομίζω ότι η επαγγελία τη θανατική ποινή είναι το αντικείμενο του ψηφίσματο και όχι η κατηγορία ει βάρο χωρομελών. Κύριε Πρέντα, νομίζω ότι είμαστε στην ίδια συνεδρίαση, αλλά φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουμε τα ίδια πράγματα. Εγώ ούτε ή άλλως είμαι ε, υπέρ ε, της χρήσης μέτρων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως, για μερικούς ε, βγάζουμε πραγματικά τα όπλα, για άλλους όμως προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Με αυτή την έννοια είναι, ήταν καρικατούρα η συνεδρίαση που είχαμε και γι' αυτό ακριβώς εγκατέλειψα και τη συνεδρίαση. Το ξέρετε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πρέντα που θα πάρει το λόγο ως εγγεγραμμένος. Ευχαριστώ. Okay, Mr. Tano, go ahead with the blue. Ο κύριος Τάνοκ έχει μπλε κάρτα. Δεν ε, αληθεύει ότι το μίσο σας ε, είναι κατά τον ΙΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο κατά τη τρομοκρατία και όχι κατά τη θανατική ποινή. Ποτέ δεν άκουσα την ομάδα σας να καταδικάζει ε, θαντικές ε, στην Κίνα, στην Κούβα ή αλλού. Η κυρία κυρια Κύριε, ε, συνάδελφε, σας ε, παραπέμπω ε, σε όσα έχω πει και για την Κούβα και για άλλες περιπτώσεις. κοιτάξτε, δεν μπορείτε να μου δίνετε μαθήματα. Εγώ δεν λέω ότι θα προστατέψω τους ε, ε, χριστιανούς έναντι των μουσουλμάνων ή οτιδήποτε. Εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης διαβίωσης όλων των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα για το κανονικό του χρόνο ομιλίας. Κύριε Πρόεδρε, εγώ λέω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην ε, περίπτωση του κυρίου Αλ Ναχίμ Αλ Νασίρη. Του έχει απαγγελθεί, κινδυνεύει να του απαγγελθεί ε, η θανατική ποινή ε, σε αποστρατιωτικό δικαστήριο. Ο Αλ Νασίρι έχει κατηγορηθεί για πάρα πολύ σοβαρά αδικήματα, συγκεκριμένα για τρομοκρατική επίθεση κατά ενός ε, ε, αμερικανικού πλοίου και ε, στρατιωτικού πλοίου και ενός γαλλικού δεξαμενόπλου, προκαλώντας τον θάνατο πολλών ανθρώπων. Πρέπει να σας πω ότι για το ΕΛΚΕ η ισχυρή διατλαντική σχέση είναι πραγματικά προτεραιότητα όμως με την προϋπόθεση να στηρίζεται, να βασίζεται ε, σε προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μία σειρά ισχυρών αρχών και αξιών. Ε, βεβαίως ε, εμείς είμαστε κατά των τρομοκρατών και είμαι θα υπέρ ε, των θυμάτων κάθε τρομοκρατικής ενέργειας αλλά από τη μία πλευρά υπάρχουν δημοκρατίες σαν τα Ηνωμένα, ε, και δικτατορίες σαν αυτές που υπερασπίζεται η κυρία Μπλε κάρτα, κυρία. Η κυρία Αναγκόμα, τι έχετε να πείτε κύριε Πρέντα το γεγονό ότι σήμερα το πρωί στο Κοινοβούλιο, πολλοί συνάδελφοι και εγώ, ακούσαμε τον, τον κύριο Τόμα Αμαμπέρκ, τον ε, Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου τη Ευρώπη και μία ερώτηση που το ετέθηκε απάντησε ότι είχε επιβεβαίωση για τι σοβαρέ υποψίε ε, σε κρυφών κέντρων ε, κράτηση στην Πολωνία και στη Ρουμανία και ότι περιμένει να προχωρήσουν οι έρευνες. Να πω, Πρόεδρε, ότι δεν έχω καμία, κανένα μίσος, παρά μόνο θαυμασμό για τη ΣΥΠΑ, που ε, προασπίζονται το κράτος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επικράτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των τρομοκρατών των οποίων σκοπός είναι να καταχραστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ευχαριστώ, κύριε Σπρέντα. Ε, ε, Ευχαριστώ την κυρία Γκόμες γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι και εγώ λυπάμαι γιατί σε όλες αυτές τις ζητήσεις ε, δεν πιστεύετε καθόλου τη ρουμανική κυβέρνηση. σα υπενθυμίζω ότι και η Ρουμανία είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι μπορούμε να τη δείξουμε μια ελάχιστη εμπιστοσύνη. Άλλωστε οι Ρουμανικέ αρχέ δεν έκρυψαν καμία πληροφορία ε, και έδωσαν όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή του όταν ζητήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα. Εμεί είμαστε ανοιχτοί και περάστε σε όλα μα τα αεροδρόμια του Βουκαρεστίου, τη Κωνσταντσα, Έχουμε και το δορυφορικό κέντρο. Ανέκαθεν δείξαμε επιθυμία συνεργασίας και δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση, καμία απόδειξη για αυτούς τους ισχυρισμούς. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτό το παιχνίδι και αυτές τις τυχομηθίες. Δεν πιστεύετε ποτέ τις διαβεβαιώσεις της ρουμανικής κυβέρνησης. Σας υπενθυμίζω κυρία Γκόμες, η Ρουμανία είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μόνο ένα λεπτό για την απάντηση, αλλά έχουμε άλλη μία μπλε κάρτα από την κυρία Βεργιά αν την αποτέχεστε. Και θα έχετε 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε. Κυρία Βεργιά. Ε, οι παρατηρήσεις του κυρίου Πρεντά ε, περισσότερο στόχο έχουν να υπερασπίσουν τη Ρουμανία παρά να ασχοληθούν με το θέμα που σας ενδιαφέρει. Πριν από λίγο με πρόσβαλε, απέφθινε ύβριση εναντίον μου. Ποτέ, κύριε Πρέντα, ούτε εδώ ούτε πουθενά αλλού δεν υποστήριξα καμία δικτατορία σε κανένα μέρο του κόσμου. Εγώ ανέκαθεν κατήγγυλα παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου και διαπράττονταν αυτέ. Θα ήθελα λοιπόν να σα ζητήσω να ανακαλέσετε τα σχόλια ει βάρο μου και σα ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό. Σα ευχαριστώ. Η απάντησή σα, κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ. Εγώ είχα καταλάβει ότι ήταν ερώτηση η μπλε κάρτα, αλλά δεν άκουσα καμία ερώτηση. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι αθέμητο να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι δημοκρατίες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες ή τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και τις χώρες ή κοινωνίες όπου η άσκηση της εξουσίας είναι αυθαίρετη, απολυταρχική, ολοκληρωτική, καταχρηστική. Δεν μπορούμε όλα να τα αντιμετωπίζουμε σαν να είναι ίσα και όμοια. Αυτά ήθελα να πω. Και αν η κυρία Βερζία αισθάνθηκε ε, προσβεβλημένη από τις παρατηρήσεις μου, λυπούμε και λυπούμε για αυτό το περιστατικό. Σας ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε το ψήφισμα. Δεν ξέρω αν θα το ψηφίσουμε άμεσα, αλλά εν περιπτώσει κάποια στιγμή θα το ψηφίσουμε μετά από την συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι ουσιαστικά αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του τι σημαίνει να είμαστε συνεπείς με τις αρχές μας και με τις αξίες μας. Γιατί το Κοινοβούλιο αυτό έχει εκφραστεί σε διάφορες περιστάσεις κατά της θαντικής ποινής, οπουδήποτε και αν λαμβάνει χώρα. Επίσης, και για το τι σημαίνει σωστή εφαρμογή του δικαίου. Αυτά τα δύο ανθρωπίνα δικαιώματα είναι δικαιώματα τα οποία εμπλέκονται στην περίπτωση Άλνα Σύρη, γιατί η σωστή απονομή δικαιοσύνη αποκλεί τι στρατιωτικέ επιτροπέ και ήδη επικρίνουμε το σύστημα, καθότι αποτυγχάνει από κάθε άποψη και δεν πληρεί τα διεθνή πρότυπα για τη δίκαια δίκη. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Σαουδάραβας αυτός αντιμετωπίζει θανατική καταδίκη από μια στρατιωτική επιτροπή, παρά το γεγονό από το 2009 ζητήθηκε από τις ε, ΗΠΑ συγκεκριμένα να μην γίνονται τέτοιες διώξεις και θαντικές καταδίκες από στρατιωτικές επιτροπές. Είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία χωρί όμω κανένα μία υποχώρηση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. you, Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Επιτροπέ Βερτίνγκερ. Η τρέχουσα κυβέρνηση τον είπα, είχε αποφανθεί στην αρχή ότι θα κλείσει το στρατόπεδο του Γκαντάναμο. Δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν αυτές οι υποσχέσεις και έτσι δεν έχουν δερματιστεί και οι στρατιωτικές επιτροπές γιατί δεν πληρούν καθόλου τα πρότυπα για την δίκαια δίκη και είναι πολύ δραματικό τώρα το γεγονός ότι μιλάμε για μια εκτέλεση πλέον, μια θαντική καταδίκη. Γι' αυτό λοιπόν το ψήφισμά μας ζητά από όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και από τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να μην εκτελεστεί ο Αλ Ασύρη. Επίσης ζητούμε να γίνει μορατόρια από πλευρά των ΗΠΑ για την θανατική καταδίκη. Και σήμερα να γνωριστεί ότι υπάρχουν 16 κράτη-μέλη τα οποία έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή και τα κράτη τα οποία εξακολουθούν να την εφαρμόζω είναι πλέον στον αριθμό 58. Ο κύριος Άλνα Σύρη κρατήτο στην Πολωνία σε μια φυλακή της CIA και πέρασε από σοβαρά βασανιστήρια. Αποτελεί αυτό ευθύνη και δική μας ε, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα βασανιστήρια. Και αν αυτό δεν το διατρανώσουμε, αν δεν αναγνωρίσουμε την ευθύνη μας, ε, αυτό δεν επιτρέπεται και η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει ότι δεν μπορούμε επιφανειακά να κατηγορούμε για αντιαμερικανισμό ή για ευρωπαϊσμό. Όχι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά γεγονότα. Και εδώ θα ήθελα να υποδείξω σε αυτά που είπε η κυρία Γκόμες, αλλά και σε αυτά που ακούσαμε στην Επιτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων, ότι πλέον υπάρχουν αποδεκτικά στοιχεία για την ύπαρξη των φυλακών αυτών στην Πολωνία. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ακούσουμε τους ε, ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Καταρχάς, ο κύριος Πόσαλτ, εξ του ΕΛΚ. Η ΕΠΑ δεν είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία, όπως αναφέρθηκε, αλλά η τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη. Αλλά δεν θα προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι η δεύτερη μεγαλύτερη δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ σε ένα τόσο σοβαρό θέμα ε, έχει εσωτερικό διχασμό. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και δικαίως αναφέρθηκε ότι η ιατρική μας σχέση με, την, ε, με τη ΣΥΠΑ βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αγωνιζόμαστε για το δίκαιο, ε, το διεθνές δίκαιο και το Γκουαντάναμο δεν συνάδει με αυτό το διεθνές δίκαιο δεν είναι μια ζώνη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε κατά των σχετικών ε, δικαστηρίων. Είμαστε υπέρ του κράτους δικαίου. Είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία δεν συνάδουν με τη θεαντική καταδική και αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία παραβιάζονται στον Κουαντάναμο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε στο σημαντικό μα σύμμαχο ότι είπα, ότι δεν αποδεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να την αποδεχτούμε και αυτό εξ αρχή ε, ήταν η θέση όλων των ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η στάση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο ότι θα πρέπει να κλείσει το Κουαντάναμο και ότι ακόμα και οι τρομοκράτε έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και ότι προ το συμφέρον των θυμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την δίκαιη τιμωρία τους. Και διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ. Και τώρα έχουμε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Τάνοκ. Την αποτέχεστε, την μπλε κάρτα κύριε Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, σέβομαι απόλυτα τον Μπέρν Πόσελτ. Για μένα η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου είναι η Ινδία. Ποτέ όμως δεν άκουσα να, να περιγράφει κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρα όπως η ΕΠΑ, η Ινδία, οι πραγματικές μεγάλες δημοκρατίες του κόσμου. Κύριε Πόσελτ, έχετε το λόγο. Ο Winston Churchill είχε πει ότι θα πρέπει να ιδρύσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης. Ο κύριος Παλέτσκης εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Η ισχύ της θανατικής ποινή ε, στις ΗΠΑ και η κατάσταση στη βάση του Γαντάναμο υπονομεύει τη θέση των ΗΠΑ Πολιτείων ως σημαντικού εταίρου για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαίρομαι για την αρχική πρόθεση του Πρόεδρου Ομπάμα να κλείσει τη βάση Γουαντάναμο, αλλά περιμένουμε μετά τα λόγια και τα έργα και την ανάληψη δράση για τη μεταρρύθμιση του συστήματο αντιμετώπιση των κρατουμένων, ιδιαίτερα στην περίπτωση της υπόθεσης Αμπτελεραχήμ Αλνασίρη. Είναι αδύνατον να εξηγήσουμε στους πολίτες της Ευρώπης ή του, του κόσμου γιατί η Ρωσία, η Ουκρανία, το Αζερβαϊτζάν ε, στην Ευρώπη ε, έχει καταργηθεί θανατική ποινή και παρόλα αυτά εξακολουθεί η ποινή αυτή να ισχύει στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ελπίζω να μην καθυστερήσουν οι χαρμόσυνες ειδήσει ε, από, την, ε, από τις Ηνωμένε Πολιτείε ως προς την κατεύθυνση αυτή. Κυρία Σάκε, από τους Φιλελεύθερους και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Κανεί δεν θα διαφωνήσει ότι η τρομοκρατία θα πρέπει να αποτραπεί και ότι οι υπόπτοι θα πρέπει να περάσουν από δίκη και να δημιουργηθούν, να προσαχθούν σε μια δίκαιη δίκη. Αλλά στον πόλεμο κατά τη τρομοκρατίας ε, διακυβεύονται ακριβώ αυτέ οι αξίε τι οποίε υποτίθεται ότι προασπιζόμαστε από την τρομοκρατία. Αν επιτρέψουμε να συμβεί αυτή η διάβρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα επιτρέψουμε στου τρομοκρατέ να νικήσουν. Αν δράσουμε με άδικο τρόπο θα αποδυναμωθούμε ακόμα περισσότερο. Η διακήρυξη του τέλους ε, της, ε, του πολέμου κατά της τρομοκρατίας ήταν ένα από τα πρώτα, μία από τις πρώτες διακηρύξεις του Πρόεδρου Ομπάμα. Ωστόσο θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη. Δεν δεχόμαστε να ε, υποδεχτούμε τους κρατούμενους στον κατάναμο και δεν παραδεχόμαστε βασανιστήρια σε ευρωπαϊκό έδαφο. Ναι, πρέπει να πληρούμε τα υψηλά πρότυπα και να ανοίξουμε αυτέ τι σκοτεινέ σελίδε τη πρόσφατη ε, ευρωπαϊκή ιστορία. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τι εμπλεκόμενε χώρε. Και αυτό φαίνεται ότι είναι δύσκολο ακόμα και για το κοινοβούλιο αυτό. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις ε, κατεπίγουσε απειλέ σε αυτόν τον κόσμο. Συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την απειλή της θραντικής καταδίκης και δεν θα πρέπει η φωνή μας να καταστεί λιγότερο ηχηρή σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να αποτελούμε ένα παράδειγμα στον ελεύθερο κόσμο σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για εχθρούς ή φίλους μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ κυρία και η κυρία Άουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Μου υπενθύμησαν συνάδελφοι ότι η σκέψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται στην καθολική εφαρμογή της προστασίας των δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα δικήματα είτε συμβαίνουν εντός είτε εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έφτασε η ώρα κατά την άποψή μου που το Κοινοβούλιο να ρίξει μια δεύτερη ε, ματιά ε, για την ενδεχόμενη εμπλοκή κάποιων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε αυτές τις παράνομες φυλακίσεις εντός της ε, ενουσιακής επικράτειας. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να πέσει φως στην ε, ε, συζήτηση αυτή έτσι ώστε να αποσαφινιστούν καταστάσεις και να αρθούν υποψίες. Σήμερα το πρωί ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Τόμος Άβερμε και του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον οποίο θαυμάζω πολύ και σέβομαι, μας είπε ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, ότι συνεχίζεται, συνεχίζονται και οι έρευνες και ότι επιθυμεί και ελπίζει στην συνέχιση της εργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μέρφη εξ ονόματος ε, της Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η υποκρισία των υπεριαλιστικών ε, ε, δυνάμεων με πολύ γλαφυρό τρόπο αποδεικνύεται στο, στην κατάσταση στον κόλπο του Γουαντάναμο βλέπουμε και ξέρουμε ποιες είναι οι ε, πραγματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί, τα βασανιστήρια, το μαρτύριο του εικονικού πνιγμού, η παράνομη κράτηση ανθρώπων στον Κουαντάναμο χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, όλα αυτά ξέρουμε ότι συμβαίνουν. Ο πρόεδρος Ομπάμα πολλά είπε, πολλές υποσχέσεις έδωσε προεκλογικά για το κλείσιμο αυτής της απεχθούς φυλακής πιστεύουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει αμέσως το Γουαντάναμο, θα πρέπει όλοι οι εκεί φυλακισμένοι και κρατούμενοι να έχουν δικαίωμα στην δίκαιη λύση, ε, θα πρέπει να λήξει η δυνατότητα χρήσης των Ιρλανδικών αεροδρομίων για παράνομη κράτηση ε, της ε, CIA και αυτό να γίνει άμεσα. Μπλε κάρτα από τον κύριο Πρέντα, παρακαλώ. Τη δέχεστε, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μέρφη εάν μπορεί με τον ίδιο τρόπο ε, ε, μπορεί να μας πει ε, και το ίδιο γρήγορα εάν βασανίζονται με αυτόν τον τρόπο και οι έγκλειστοι στις φυλακές της Κούβας. Κύριε Μέρφη, παρακαλώ. Όπως και η κυρία Βερζιά προηγουμένως ε, είπε, ε, λέω και εγώ ότι δεν δέχομαι την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οπουδήποτε και αν λαμβάνει η χώρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω πάντως ότι μιλάμε για τον κόλπο του Γκουαντάναμο, μιλάμε για μυστικές ε, φυλακές, μιλάμε για χρήση παράνομων διαδικασιών από τις ΗΠΑ και αυτό θα πρέπει να καταδικαστεί εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος but Ας μην χάνουμε την προοπτική εδώ. Έχουμε 775 κρατούμενους από τότε που άνοιξε το Γουαντάναμο, η βάση του Γουαντάναμο. Μέσα στο, στην αίθουσα αυτή θα μπορούσαν να χωρέσουν οι 775 κρατούμενοι που κρατήθηκαν από την αρχή της λειτουργίας βάσης του, του, κρατη, της φυλακής του Γουαντάναμο. Εμεί ενδιαφερόμαστε φυσικά για τι ε, δημόσιε ελευθερίε και για το κράτος δικαίου, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένοι κρατούμενοι όντως ε, έχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, είχαμε ένα Βρετανό υπήκο που συνελήφθη στο Αφγανιστάν με όπλα ε, αποδεδειγμένο μέλος του, του, των Ταλιμπάν εξήγησε ότι βρέθηκε στο Αφγανιστάν για να παρακολουθήσει μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών παρόλο που βρέθηκε με όπλα ε, φυσικά θέλουμε να ε, δούμε την ε, νομική διαδικασία που ισχύει για το Γουαντάναμο, αλλά το θέμα της, των δημοσίων ελευθεριών στον κόσμο θα αντιμετωπίζονται καλύτερα αν το Κοινοβούλιο ενδιαφερόταν περισσότερο για τις επιχειρήσεις ότι αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης σε μεγάλο βαθμό από τη φύση του παραβιάζει τις, ε, τα νομικά εχέγγυα ε, κατά των αυθαίρετων κρατήσεων. Και πάνω από ένα εκατομμύριο υπόκειται σε αυτόν τον κίνδυνο, που είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός και πιο εντυπωσιακό από τους 775 κρατούμενους στο Βαντάναμο. Ο κύριος Σιλβέστρης. Κύριε Πρόεδρε, πέντε μέρες πριν μάθαμε ότι επισήμως ε, απεγγέλθηκαν κατηγορίες σε πέντε που θεωρούνται ύποπτοι για τις επιθέσεις του Δήμου Πύργου ε, ε, Θα, διοργανωθεί από ό,τι φαίνεται δίκη για αυτούς τους τρομοκράτες ενώπιον στρατιωτικού δικαστηρίου. Παρόλα αυτά και πρέπει πρώτα απ' όλα να καταδικάσουμε βεβαίως τις τρομοκρατικές ενέργειες. Όμω θα πρέπει ταυτοχρόνω να πούμε ότι θα πρέπει να ε, να σταματήσει η θανατική ποινή για, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και για οποιοδήποτε έγκλημα. Επίση, ότι θα πρέπει να καταγγέλουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οποτεδήποτε και οπουδήποτε ε, γίνονται ε, αυτά. Ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να θυμίσουμε και στους συναδέλφους της ΓΚΟΕ ότι το τελευταίο γραφείο Ζαχάροφ δεν ε, ήθελα να δοθεί γιατί θεωρούσαν ότι είναι εγχειρηματοποίηση του βραβείου. Ο κύριος Ζακένα, πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αρνούμαστε να καταδικάζουμε, να καταδικάσουμε τη ΣΥΠΑ για την εγκληματική τους συμπεριφορά στο Γουαντάναμο και αρνούμαστε την ευθύνη χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ επέτρεψαν την φυλάκιση κρατουμένων και τα βασανιστήρια σε μυστικέ φυλακέ τη ε, CIA στο έδαφο τη. Είχαμε παιδιά στρατιώτε που συνελήφθησαν και βασανίστηκαν στο Γουαντάναμο κατά παράβαση τη σύμβαση τη UNICEF. Ε, πώς ε, άλλες φορές καταδικάζουμε ε, κάποιες δικτατορίες και επιβάλλουμε κυρώσει όταν ε, μιλούμε για τη ΣΥΠΑ δεν ε, ε, είμαστε εξίσου αυστηροί. Είναι οικουμενικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους ε, πολίτες του κόσμου. Θα πρέπει και, να, και τη είπα να τις δικάσουμε για, τα, για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τις συνένοχες με τη ΣΥΠΑ χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο και να τεθεί τέρμα στο βασανισμό και στη θανάτωση στο όνομα του αντιτρομοκρατικού αγώνα. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να επαναλάβουμε τις εκκλήσεις μας για κλείσιμο της βάσης του Γουαντάναμο και επαναφοράς ε, της περιοχής αυτής στην Κούβα για να αποκαταστήσει την ακεραιότητα της εδαφικής της επικράτειας. Ε, ε, Συνάδελφοι, όπως και το δικαίωμα στη ζωή είναι ένα πολύ ιδιαίτερο δικαίωμα μεταξύ των ανθρωπινών δικαιωμάτων, η θανατική καταδίκη δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η Ευρώπη του σήμερα αποτελεί μοναδική, τη μοναδική περιοχή του κόσμου όπου δεν έχει θέση η θανατική ποινή. Με λυπηρό παράδειγμα, με λυπηρή εξαίρεση την ε, Λευκορωσία. Είμαι υπέρ της κατάργησης της θανατικής καταδίκης παντού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διατλαντική σχέση είναι πραγματικά ανεκτήμητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η αμοιβαία μας συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να υποστηρίξω την έκκληση στις αρχές των ΗΠΑ να μην επιβάλλουν την θανατική καταδίκη στην περίπτωση του Αλ Νασίρη. Συνοψίζοντας, Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που καλούν τις χώρες που εξακολουθούν να εφαρμόζουν την θανατική ποινή να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο και να καταργήσουν την θανατική ποινή και να καταστεί αυτό μια καθολική αξία. Όλες οι εκτελέσεις όπου και αν λαμβάνουν χώρα θα πρέπει να καταδικάζονται. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Κούκα. Κύριε Κρέτσου. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες που είπαν ότι όταν εξακοντίζονται σοβαρές κατηγορίες κατά μιας χώρας, να μην γίνεται αυτά βασάνιστα, να στηρίζονται από βάσιμες αποδείξεις. Δεν είναι θέμα διπλών μέτρων και σταθμών, είναι θέμα αξιοπιστίας. Φυσικά όλες οι χώρες έχουν το ηθικό καθήκον να καταργήσουν τη θανατική ποινή. Οι διατλαντικέ σχέσεις στηρίζονται σε κοινέ αξίε και αρχές και ευελπιστώ ότι οι αμερικανικές αρχές ε, θα ε, εισακούσουν το αίτημά μας για την κατάργηση τη θανατική ποινή. Θα ήθελα να απαντήσω στο συνάδελφο Πρέντα και να του πω ότι η θέση μας για τη θανατική ποινή δεν σημαίνει ότι υποτιμούμε τη στρατηγική μας σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε μια, με ανώτερης ποιότητας εταιρική σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο για το ΕΛΚ προτεραιότητα η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τους σοσιαλιστές είναι επίσης προτεραιότητα. Κύριε Πρέντα, στο διαδικασία του Catch the Eye δεν προβλέπεται μπλε κάρτα. Είχατε προηγουμένως αρκετό χρόνο για να μιλήσετε. κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα. Θα ήθελα... Θα ήθελα να τονίσω την περίπτωση του Αλνασάρη. Είναι βληματική όχι μόνο λόγω του Γαντάναμο και της ανατικής ποινής, αλλά και επειδή αποτελεί έναν από τα, ένα από τους δύο κρατούμενους σε κέντρα ε, κράτηση στην Ευρώπη, μαζί με τον Αμπού Σουμπάκη και ελπίζουμε ότι η διαδικασία απόδοσης της δικαιοσύνης θα επιταχυνθεί στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το τελικό ψήφισμα να περιλαμβάνει σαφή έκκληση για αποτελεσματικές έρευνες στην συνενοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των, τα σχετικά προγράμματα. Ωστόσο, είναι σημαντικό αυτό να συνδυαστεί με μία έκθεση που ε, συμφώνησε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να συμπεριληφθεί και σε μια νέα έκθεση πρωτοβουλίας. Και φαίνεται ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το ζήτημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα. Ο κύριος Φεραίρα. Κύριε Πρόεδρε, Έχουμε ένα άλλο λυπηρό παράδειγμα της πολιτικής διπλών μέτρων και σταθμών, που είναι συνηθισμένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ μιλούμε για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρου των Αμερικανικών αρχών, αυθαίρετες και απαράνομες κρατήσεις, καταστρατήγηση του δικαιώματος δικής δίκης, εφαρμογή βασανιστήριων, απαγγελία θανατικής ποινής και μάλιστα τέτοιες παραβιάσεις πολλές φορές έγιναν με τη συνενοχή χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραχώρησαν το έδαφος, της, το έδαφος του CIA για τις παράνομες δραστηριότητές της. Δεν μιλάμε τίποτα όμως για καταδίκη των Αμερικανικών αρχών, δεν μιλούμε τίποτα για καταδίκη των χωρών που συνεργάστηκαν μαζί τους. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτήσει μετατράπηκαν σε αιτήματα. Στο πρώτο σημείο της, του ψηφίσματος μιλούμε για την ενίσχυση της διατλαντικής σχέσης που στηρίζεται σε κοινέ αρχές και αξίες με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πού είναι αυτός ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λυπηρό κάτι τέτοιο. Γιατί πέραν της έκκλησης να κλείσει η βάση του Γουαντάναμο, πιο σημαντικό θα ήταν να ανακτήσει η Κούβα την κυριαρχία σε αυτό το τμήμα της ε, επικράτειά τη που παράνομα κατέχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Σα ευχαριστώ το λόγο κυρία Κορχόλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα συμφωνούμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει στον αντιτρομοκρατικό αγώνα σε συνεργασία με τους εταίρους της. Βέβαια, ο αντιτρομοκρατικός αγώνας δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν κατά της θανατικής ποινής και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του κυρίου Αλνασίρη. Έχουμε αφενός την ανάγκη κατάργησης της θανατικής ποινής αλλά απ' την άλλη έχουμε και την ανάγκη καταπολέμησης των αιτίων της τρομοκρατίας. Οι διατηλαντικές σχέσεις στηρίζονται σε κοινέ αξίες που είναι οι οικουμενικές αξίες της ισότητας μπροστά στη δικαιοσύνη, της δημοκρατίας κτλ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να κλείσουν το Γουατάναμο, να καταργήσουν τις στρατιωτικές επιτροπές και να πράξουν τα δέοντα στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Δύο ακόμη ομιλητές. Ο κύριος Κατσμάρεκ πρώτα οι τελευταίοι ομιλητέ, το ΚΑΤΣΔΙ. Κύριε Πρόεδρε, πολλοί ευρωβουλευτέ μίλησαν για αποδείξει ό,τι αφορά την ύπαρξη φυλακών στην Ρουμανία και την Πολωνία και μυστικές φυλακές όπου διαπράχθησαν ε, βασανιστήρια. Παρακαλώ αυτές τις αποδείξεις που έχετε να τις στείλετε στην εισαγγελία της Πολωνίας γιατί στην Πολωνία η δικαστική αρχή είναι ανεξάρτητη από την κυβέρνηση και μάλιστα ε, την κατάσταση την παρακολουθούν ε, το Συμβούλιο της, του Ελσίνκη. Αν έχετε τέτοιε αποδείξει για τι δύο περιπτώσει που μα είπατε, γιατί δεν τι επιδίδετε στην εισαγγελική αρχή τη Πολωνία για να διερευνήσει αυτέ τι αποδείξει και του ισχυρισμού. Και μάλιστα είχαμε και ειδική επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Ένα από τα μέλη τη Επιτροπή σήμερα είπε στην Πολωνία ότι υπάρχουν γραπτέ αποδείξει ε, με υπογραφή του προηγούμενου σοσιαλιστή ε, πρωθυπουργού που μίλησε για το θέμα της, ε, των μυστικών φυλακών ε, όταν το ρώτησα, είδατε με τα μάτια σε αυτό το έγγραφο, μου είπε ο βουλευτή, δεν το είδα με τα μάτια μου, αλλά άκουσα ότι υπάρχει. Το θέμα είναι όχι μόνο να μεταφέρουν κάποιοι φημολογίε, να είναι αυτό τι μάρτυρε και να, αν έχουν στοιχεία και αποδείξει, να τι δώσουν στην εισαγγελία. Η επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Αυτή η συζήτηση εν μέρη και η πολιτική αντιπαράθεση εδώ ίσως να μην ε, εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτού του ψηφίσματος παρά το γεγονός ότι εδώ στην αίθουσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να προσπίσουμε το δικαίωμα του κάθε πολίτη τα δικαίωμα για μια δίκη και είμαστε ασφαλώς και κατά της αντικής καταδίκης. Παντού και ανεξάρτητα από τα εγκλήματα τα οποία αφορούν οι καταδίκες. Οι κατηγορίες ε, κατά του Αλνασίρη είναι πολύ μεγάλες, κατηγορείται για μεγάλα εγκλήματα και θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν αποδεχόμαστε τις πράξεις του, δεν αποδεχόμαστε την τρομοκρατία, αλλά θέλουμε να προασπιστούμε το δικαίωμα κάθε ανθρώπου για μια δίκαιη δίκη και είμαστε επίσης υπέρ τη συνολική κατάργηση τη αντικής καταδική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα ήρθε η ώρα για την Επιτροπή και τον Επιτρόπο την λέει ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ στον αγώνα κατά τη τρομοκρατία. Ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη η αξία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμα και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τον Ιούνιο του περασμένου έτους εμείς και η ΕΠΑ προβήκαμε σε μια κοινή διακήρυξη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας όπου αναφέρεται ότι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συμφωνία προβλέπει όλες οι δίκες να γίνονται σε ένα νόμιμο πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη δίκαιη δίκη και σε όποιο βαθμό γίνεται θα διασφαλίζει μια διαφανή διαδικασία. Εδώ και πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά να κλείσει το στρατόπεδο στο Γκουαντάναμο. Θεωρούμε ότι η μακρά κράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ομπάμα πριν από δύο χρόνια ανακοίνωσε το κλείσιμο του Γκαντάναμο εντός ενός έτους και μάλιστα την διέταξε. Ε, συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ επί ενός πλαισίου για την υποδοχή κάποιων κρατουμένων. Είμαστε επίσης ε, πρόθυμοι να συνεργαστούμε στενά με τη ΣΥΠΑ σε περίπτωση που θα κλείσει τον Κουαντάναμο. Παρά του διατάγματος του Μαρτίου του Προέδρου με την οποία ε, εγκρίθηκε η κράτηση κάποιων ατόμων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα ληφθεί η απόφαση να, κλειστεί, να ε, κλείσει το συντομότερο δυνατόν το στρατόπεδο κράτηση. Η στάση μα είναι σαφή. Απορρίπτουμε την θανατική καταδίκη υπό όλε τι συνθήκε. Αυτό ισχύει για όλες τι χώρες του κόσμου. Καλούμε λοιπόν ρητά της ΕΠΑ να καταργήσουν την θανατική ποινή σε όλη την επικράτεια της χώρας και σε όλες τις πολιτείες ε, της, ε, των ΕΠΑ. Και γι' αυτό λοιπόν ανησυχούμε για τους κρατούμενους εκείνους στους οποίους ε, απειλείται, οι οποίοι απειλούνται με την θαντική καταδική. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί αν ο Αλ και οι πέντε συνένοχοι του στις τρομοκρατικές εμ, ενέργειες θα μπορούσαν να καταδικαστούν σε θάνατο. Να σας διαβεβαιώσω ότι μου παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μας απασχολεί το κατά πόσο είναι δίκαιη η δίκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε πίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το Γουαντάναμο. Η ψηφοφορία θα γίνει αμέσως μετά το πέρας της συζήτησης και του επόμενου σημείου που αφορά την Ουκρανία και την υπόθεση της Γιούλιας Τιμοσέγκο και άλλων μελών